Please, does everybody his voting card? Έχουν όλοι την ε, κάρτα για την ηλεκτρονική ψηφοφορία, λέει η πρόεδρος. Αλλιώς να αναβάλουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία, τόσο ώστε να μπορεί ο καθένας να πάει να ψάξει την κάρτα. Απλώς πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι πρέπει να έχετε την κάρτα σας. Guten Morgen. Ich bedanke mich beim Kollegen äh, Suoni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 nevealov zu dem thema jugend. ich bitte nevealov das wort zu nehmen. bitte. Ďakujem vám pekne. Prajem všetkým dobré ráno. Ευχαριστώ. Να είμαι σύντομη για να πάμε στις ψηφορίες. Το 2010 ήταν η χρονιά για την καταπολέμηση της ε, φτώχειας του κοινού αποκλεισμού αλλά τελικά εκτός από τους ηλικιωμένους και είναι, είναι ευάλωτη η κοινωνική ομάδα. Γι' αυτό και χαιρόμαστε που το Κοινοβούλιο διάλεξε να ασχοληθεί με αυτό το θέμα και το τι κάνουν οι νέοι στην ε, αγορά εργασίας. Οι νέοι μόλις ε, τελειώσουν την ε, ε, εκπαίδευσή τους, τον κύκλο της παιδείας, ε, την, την βγουν από το πανεπιστήμιο. Έχουμε το 21% των νέων οι οποίοι δεν έχουν δουλειά. Η έκθεση αυτή προέρχεται από την Επιτροπή Απασχόλησης. Κάτι γνώμη μου είναι πάρα πολύ αξιόλογη και αφορά συγκεκριμένα διαβήματα, συγκεκριμένες ε, πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να έχουμε κάποια νέα στήριξη, κέντρα στήριξη για τους νέους και έτσι να γίνει πιο εύκολη η πρόσβαση του αγορά εργασία. Παιδεία και κατάρτιση αναφέρονται στην έκθεση. αυτή που πρέπει να εξετάσει η Επιτροπή μα που θα αφορά επομένω την εκπαίδευση των νέων, την επαγγελματική του κατάρτιση, κάποιες εξειδικευμένες γνώσεις πρέπει να αποκτήσουν. Άλλωστε είναι η υπόθεσή μας και η παιδεία, αλλά και η ισόβια κατάρτιση. Θα πρέπει επομένω, όσο γίνεται περισσότεροι νέοι, να μπορούν να αποκτήσουν όσο γίνεται περισσότερα προσόντα γιατί το πρόβλημα δεν είναι τα πανεπιστημιακά πτυχία, είναι το να βρουν μια δουλειά μόλι τελειώσουν τι σπουδέ του. Επομένω, αυτό χρειάζεται. Μόλι κανεί τελειώσει τι σπουδέ, να μπορεί να αποκτήσει κατόπιν κάποιε άλλε γνώσει σε κάποια σχολή, σε κάποιο άλλο πανεπιστήμιο. Και σας υποβάλλω το κείμενό μου, φαντάζομαι ότι ήδη έχετε ρίξει μια ματιά, δεν είναι και πολύ μεγάλο το κείμενο αυτό. και θα συναντηθούμε αργότερα με τους και ηγητές για να δούμε πώς όλες σας τις ε, παρατηρήσεις θα μπορούμε να συντάξουμε στο κείμενο. Ευχαριστώ. Μπαδιά Κουτσέτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Νεβεντάλοβα για την ε, έκθεσή της. Είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά τα οποία λέει, είναι πολύ εύστοχα. στην έκθεση που πρόκειται από την ε, Επιτροπή Απασχόλησης. Ίσως πρέπει να πούμε κάτι για την διαδικασία της ε, Μπολόνια γιατί έτσι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ιδέες που κατεβάζει η κυρία Νεβεντάλαβα γιατί είναι νομίζω η εκθεσιστεί κάτι που χρειαζόταν και είναι πάρα πολύ σωστή. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και να πω στην κυρία Ντελούκα ότι ίσως το θέμα των ξένων γλωστών πρέπει να είναι λίγο πιο σαφές και να τονιστεί περισσότερο. Διότι ξένες γλώσσες ε, όταν πρόκειται για πρακτική κατάρτιση είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που γίνεται στο γυμνάσιο στο θέμα αυτό λοιπόν στις ξένες γλώσσες θα πρέπει να εστιαστούμε περισσότερο στην εργασία κατά τρόπον ώστε οι νέοι που έχουν λιγότερο ενδιαφέρον να μάθουν γλώσσες να καταλάβουν γιατί πρέπει να τις διδαχθούν γιατί αν κάνουν μία ε, μετεκπαίδευση στο εξωτερικό και δεν γνωρίζουν ε, τους όρους της ε, δουλειάς τους διότι με την απλή εκμάθηση της γλώσσας μαθαίνουν όταν κάνουν συζήτηση. Λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο ίσω θα έπρεπε να αναφερθεί. Επίση, όταν μιλάμε για το θέμα Λεωνάρντο θα έπρεπε τουλάχιστον να το αναφέρουμε διότι το Λεωνάρντο είναι που ειδικεύεται στον τομέα αυτό και ο Έρασμος. Ο Έρασμος, το πρόγραμμα Έρασμος έχει αναλάβει το πρόγραμμα για τους φοιτητές. Παλιά όλα αυτά ήταν στο πρόγραμμα Λεωνάρντο, τώρα είναι στο πρόγραμμα Οπότε ίσως θα έπρεπε να αναφερθεί για να είναι πλήρης η εικόνα. Υπάρχει κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι, γιατί είχε προβλεφθεί ότι αυτό θα γίνει στο τέλος. Οπότε ε, ε, δεν, ε, ε, δεν επιπλήττω κανέναν. Θέλαμε απλούστατα να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο μέχρι ότου να έρθουν τα μέλη της Επιτροπής με τις κάρτες ψήφου. Ψηφοφορία. Θέλει κάποιος άλλος κάτι να προσθέσει. Ε, ευχαριστώ. Όσον αφορά την διαδικασία της Μπολόνια θα πρέπει να αναφερθεί ε, και για τις ξένες γλώσσες ε, πρέπει να πάρουμε το παράδειγμα της Σουηδίας που μου αρέσει διότι ε, περιλαμβάνονται οι ξένες γλώσσες στο τυποποιημένο πρόγραμμα εκμαθής διδασκαλίας. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι καλύτερο. Ευχαριστώ. Ωραία. Λοιπόν, να σας πω ότι μέχρι την Πέμπτη στις 25 Μαρτίου 12 το μεσημέρι θα έχουμε, ε, θα έχουμε την προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Αυτή την εβδομάδα δηλαδή. Και έτσι ολοκλήρωσα. Ε, θα δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφο Σόνικ. Ερχόμαστε... Όχι, ε, λάθος θα ε, ψηφίσουμε πρώτα την έκθεση Carl Σμιτ, Πάλ Σμιτ, Διάλογος Πανεπιστημίων Επιχειρήσεων. Μια νέα εταιρική σχέση για τον εξυγχωρισμό των Πανεπιστημίων της Ευρώπης. Η έκθεση αυτή είχε παρουσιαστεί στις 23 Φεβρουαρίου, μετά η προθεσμία υποβολής τροπολογιών ήταν μέχρι 1η Μαρτίου και είχαμε 109 τροπολογίες. Έχουμε και μια γνωμοδότηση από την Επιτροπή Ήτρε και γι' αυτό θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Σμιτ εάν θέλει κάτι να προσθέσει πριν την ψηφοφορία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου αναθέσατε αυτή την έκθεση που μου δίδαξε πολλά. Δηλαδή ότι και στην Ουγγαρία έχουμε πολλά προβλήματα για τους νέους ακαδημαϊκούς οι οποίοι βγαίνουν από τα πανεπιστήμια και ψάχνουν δουλειά και δυσκολεύονται να την ε, επιτύχουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους επιπλέον για όλες αυτές τις τροπολογίες και στη ρήτα. θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ωραία. Τότε αρχίζουμε την ψηφοφορία. Όπως σας είχα πει από την αρχή θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Έχετε όλοι τις κάρτες σας. Παράγραφος 1, τροπολογία 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ ψηφίζεται μάλλον ηλεκτρονικά απορρίπτεται. Δεν χρειάζεται κάθε φορά να σας λέω τους αριθμούς διότι τους βλέπετε ε, στις οθόνες. Τροπολογία Ήτρε. Αρχίζει ψηφοφορία, λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ήτρε δύο, αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη εγκρίνεται. Ήτρε 3. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. Παράγραφος 1α 18. Ε, Αρχίζει. Λίγη. Απορρίπτεται. 19. Άρχεται ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. 20. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 21. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 22. Εγκρίν, ε, ξεκινά. Λίγη. Απορρίπτεται. 23. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 24. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 25. Ξεκινά. Λίγη. Απορρίπτεται. 26. Ξεκινά. Λίγη. Απορρίπτεται. 27. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 28. Αποσύρθηκε. και 29 ξεκινά ψηφοφορία. Λίγη. Ξεκινά ψηφοφορία, λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 30. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 31. Ξεκινά. Λίγη εγκρίνεται. Ήτρε 2. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. Ήτρε 16. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. Ήτρε 21. Ε, ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1 του κυρίου Βης. Ε, ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 32. Καταπίπτει. Καταπίπτει το 32. 33. Ε, ξεκινά. Λίγη. Απορρίπτεται. 34. Σε δύο τμήματα. Πρώτο μέρος ξεκινά Λίγη. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. 35. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Ε, λίγη. Εγκρίνεται. 37. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 38. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ξεκινά ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος ξεκινά. Λίγη. Απορρίπτεται. 39. Ξεκινά. Λίγη εγκρίνεται 40 αποσύρεται και το 41 42 σε δύο μέρη ξεκινά στο πρώτο μέρος κλείνει εγκρίνεται δεύτερο μέρος ξεκινά λίγη εγκρίνεται 43 Μάλλον το δεύτερο μέρος απορρίπτει και με συγχωρείτε λέει η πρόεδρος απερίφθη. 43 ε, ξεκινά, λίγη, απορρίπτεται. 44 ξεκινά, λίγη, απορρίπτεται. 45 ξεκινά, λίγη, εγκρίνεται. 46 ξεκινά, λίγη, εγκρίνεται. 47 ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 48 ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 49. Δεν δουλεύει το μηχάνημά σας. Επαναλαμβάνουμε το 48. Ξεκινά. Δουλεύει τώρα. Λίγη. Εγκρίνεται. 49. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 50 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος ξεκινά ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. 51 ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 52. Ξεκινά. Λίγη. Απορρίπτεται. 53. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 54. Ξεκινά. Λίγη. Απορρίπτεται. 55. Ξεκινά. Λίγη εγκρίνεται 56 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 58 ξεκινά λίγη εγκρίνεται Ήτρε 10 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 59 ξεκινά λίγη εγκρίνεται Λοιπόν, θα σα λέω ανοίγει και κλείνει, ε, να πηγαίνουμε πιο γρήγορα. 61 ε, ανοίγει, κλείνει. Επαναλαμβάνουμε. 61 ξεκινά, λίγη. Εγκρίνεται. 62 ξεκινά, λίγη. Εγκρίνεται. 63 ξεκινά, λίγη απορρίπτεται 64 αποσύρεται 65 ξεκινά λίγη 65 ξεκινά λίγη απορρίπτεται 66 ξεκινά λίγη απορρίπτεται 67 ξεκινά Κλείν, ε, λίγη. Απορρίπτεται. 68 ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 69 ξεκινά. Λίγη. Απορρίπτεται. Ήτρε 7 ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 70 ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται απορρίπτεται 71 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 72 ξεκινά κλείνει εγκρίνεται 74 αρχίζει τελειώνει εγκρίνεται 75 σε δύο μέρη πρώτο λίγη δεύτερο τμήμα ξεκινά Λίγη. Απορρίπτεται. 77. Ξεκινά. Λίγη. Απορρίπτεται. 78. Ξεκινά λίγη. Απορρίπτεται. 81. Ξεκινά. Λίγη. Απορρίπτεται. Ξεχάσαμε το 79. 79 με συγχωρείτε. Επανερχόμαστε στο 79. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 81 ε, τώρα. Ανοίγει, κλείνει. Απορρίπτεται. 72 ε, ξεκινά λίγη. Εγκρίνεται. 84 ε, ξεκινά. Λίγη. Απορρίπτεται. 85 ξεκινά. Λίγη εγκρίνεται 86 ξεκινά λίγη απορρίπτεται 87 ξεκινά λίγη εγκρίνεται επαναλαμβάνουμε λοιπόν την 87 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 88 ξεκινά λίγη Εγκρίνεται. 89. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 90. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 91. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. Ήτρε 8. Ανοίγει. Κλείνει. Εγκρίνεται. Ήτρε 19. Ε, αρχίζει. Λίγη. Εγκρίνεται. Ήτρε 9 εγκρίνεται 93 ξεκινά λίγη εγκρίνεται πρώτη συμβιβαστική αρχίζει λίγη πάλι δεν λειτουργεί επανερχόμαστε στην πρώτη συμβιβαστική επειδή προχωράμε πάρα πολύ γρήγορα νομίζω ότι πατάμε το κουμπί πριν ανάψει αυτό το φωτάκι. Καλύτερα να περιμένουμε να ανάψει το φωτάκι και μετά να πατήσουμε το κουμπί. Έτσι θα δουλεύει καλύτερα. Ε, λοιπόν, έχουμε ε, ε, συμβουλές από τη, τη συνάδελφο πρώτη συμβαστική ξεκινά λίγη εγκρίνεται 94 ξεκινά λίγη απερίπτεται 95 σε δύο τμήματα Πρώτο τμήμα ξεκινά, α, κλείνει, εγκρίνεται. Δύο, Ξεκινά, κλείνει, εγκρίνεται. 98. Ξεκινά, λίγη, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 100 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 101 ε, ξεκινά λίγη εγκρίνεται 103 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 104 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 106 ξεκινά λίγη Το 105 γιατί δεν το ψηφίζουμε. Το 105 δεν χρειάζεται να το να το ψηφίσουμε. Χρειάζεται. Οπότε τεχνικό λάθος. 105. 105. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. ήταν μόνο ε, μία υπόδειξη ότι εάν υιοθετηθεί θα είναι ένα εκτιμώντας και όχι τροπολογία. Ε, το 106 υπέρ ε, κλείνει, εγκρίνεται. Ήτρε 13 αρχίζει. Το 13 είναι περιττό. 107 κόστα. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 108 ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. Ένα. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. Δύο. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. Τρία. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. Τέσσερα σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ξεκινά. Λίγη εγκρίνεται δεύτερο μέρος ξεκινά κλείνει απορρίπτεται Εξι, ξεκινά κλείνει απορρίπτεται Επτά, ξεκινά λίγη εγκρίνεται Οχτώ, ξεκινά λίγη εγκρίνεται Εννέα, ξεκινά λίγη απορρίπτεται Δέκα, ξεκινά Λίγη. Απορρίπτεται. 11. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 12. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 13. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 14. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 15 ξεκινά. Λίγη απορρίπτεται 16 λίγη απορρίπτεται τώρα ήτρε Όσον αφορά τις τροπολογίες της Ήτρε που είναι στην τελευταία σελίδα, αυτές θα ενσωματωθούν στο κείμενο σύμφωνα με την, ε, τον εσωτερικό κανονισμό. Ψηφίζουμε τώρα ολόκληρο το κείμενο. Ξεκινά λίγη. Ε, ομόφωνη αποδοχή, ε, θερμία συγχαρητήρια στον εισηγητή. Η κυρία Βερζιά δεν μπορούσε να ψηφίσει, αλλά είναι και αυτή υπέρ. Α, ψηφίσατε κατά. Συγγνώμη, συγγνώμη. Λοιπόν, μία, μία ψήφος εναντίον καταψηφίζει και αυτό ομορφαίνει το όλο πράγμα. Μαρή Τερέζ, δεν μπόρεσες να ψηφίσεις. Και 29 υπέρ και μία κατά, γιατί έχουμε άλλες δύο ψήφους υπέρ. Ε, λοιπόν, να στα πρακτικά παρακαλώ. Τώρα ερχόμαστε στην επόμενη έκθεση στην έκθεση Παπα-Νικολάου, η οποία είναι ακόμη χειρότερη από πλευράς τροπολογιών. Πρέπει να σας πω ότι στην επόμενη ψηφοφορία εγώ θα φύγω, θα με αντικαταστήσει κάποιος άλλος. Μήπως να τα λέω αγγλικά θα είναι πιο απλά. Όχι. Καλά λειτουργεί και έτσι. Αγαπητέ συνάδελφε, θέλετε κάτι να πείτε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, από όλες τις συζητήσεις που έχουν γίνει στα πλαίσια της Επιτροπής μας, νομίζω έχει προκύψει το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει από όλους τους συναδέλφους. Θέλω να ευχαριστήσω για όλες τις τροπολογίες και για όλα τα σχόλια. Θέλω να ευχαριστήσω ειδικά τους συζητητές όλων των πολιτικών ομάδων, να ευχαριστήσω και τη γραμματεία μας για την πολύ στενή συνεργασία και τη συνδρομή της όλο αυτό το διάστημα. Ε, μία μόνο παρατήρηση. Αυτή η έκθεση και αυτή η πρωτοβουλία που έχει η Επιτροπή μας αυτή την περίοδο δεν σταματάει εδώ, πρέπει να συνεχιστεί. Θυμίζω ότι για τις πολιτικές για την νεολαία ε, έχουμε επικουρικότητα, άρα εμείς κάθε φορά με τις τοποθετήσεις μας, με τον διάλογο, με τα συμπεράσματά μας πρέπει να προσπαθούμε να εξηγούμε και να πείθουμε τα κράτη-μέλη ότι η δουλειά που γίνεται εδώ αξίζει να ενσωματώνεται και να αφομοιώνεται στις πολιτικές ε, κάθε κράτου μέλους προς όφελος κάθε νέου ανθρώπου σε όλη την Ευρώπη. Νομίζω αυτή η έκθεση αποτελεί την αρχή για ακόμη πιο σημαντική προσπάθεια της Επιτροπής μας στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ για όλη τη συνεργασία και πάλι ε, και ευελπιστώ ότι και στην Ολομέλεια ε, θα μπορέσουμε, θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε και περισσότερα. vielen Dank. Ωραία, ευχαριστώ. Προχωράμε στην ψηφοφορία. Παράγραφος 3. Τροπολογία 30. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 31 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 32. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. Πρώτη συμβιβαστική ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 36. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 37. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 38. Ξεκινά. Λίγη εγκρίνεται 39 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 40 ξεκινά λίγη απορρίπτεται 41 προφορική τροπολογία ξεκινά λίγη εγκρίνεται 42 αποσύρεται 43 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 44 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 45 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 46 ξεκινά λίγη απορρίπτεται 47 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 48 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 49 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 50 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 51 κλείνει εγκρίνεται 52 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 53 ξεκινά κλείνει εγκρίνεται 54 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 55 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 56 ξεκινά ε, λίγη εγκρίνεται 57 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 58 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 59 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 60 ξεκινά λίγη εγκρίνεται Β συμβιβαστική ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 63. Ξεκινά. Λίγη. Απορρίπτεται. Η 63 μιλάμε. Βεζιά μπίσκι ταβαρές. 66. Ξεκινά. Λίγη. Απορρίπτεται. 67. Ξεκινά λίγη, εγκρίνεται, 68 ξεκινά, λίγη, εγκρίνεται, 69 ξεκινά, λίγη, εγκρίνεται, 70 ξεκινά, λίγη, εγκρίνεται. Συμβαστική γιώτα ξεκινά λίγη εγκρίνεται 73 ξεκινά, λίγη, εγκρίνεται. 74 ξεκινά, λίγη, εγκρίνεται. 75 ξεκινά, λίγη, εγκρίνεται. 76 ξεκινά, λίγη, απορρίπτεται. Συμβιβαστική C. Ξεκινά, λίγη, εγκρίνεται. 77 ξεκινά, λίγη, εγκρίνεται. 80 ξεκινά λίγη, εγκρίνεται. 81 ξεκινά λίγη, εγκρίνεται. Συμβιβαστική D ξεκινά, λίγη, εγκρίνεται. 86 ξεκινά, λίγη, εγκρίνεται. Συμβιβαστική ε. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 90. Ξεκινά. Λίγη. Απορρίπτεται. 92. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 91. Ξεκινά. Λίγη. 93. Ξεκινά. Λίγη απορρίπτεται 94 ξεκινά λίγη εγκρίνεται Συμβασική F ξεκινά λίγη εγκρίνεται 97 κλείνει απορρίπτεται νομίζω απορρίπτεται 101 υπέρ κατά ε, κλείνει 102 ξεκινά κλείνει εγκρίνεται 103 ξεκινά κλείνει απορρίπτεται 104 υπέρ ε, κλείνει εγκρίνεται 106 ξεκινά κλείνει εγκρίνεται 107 ξεκινά λίγη Εγκρίνεται. 108. Ξεκινά. Κλείνει. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική G. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 113. Κλείνει. Απορρίπτεται. 114. Έχει πρώτο και δεύτερο μέρος. Το πρώτο μέρος ξεκινά, λίγη, εγκρίνεται. Δεύτερο ξεκινά, λίγη, εγκρίνεται. 115 ξεκινά, λίγη, εγκρίνεται. 117 ξεκινά. 116 με συγχωρείτε λέει πρόεδρος, ξεκινά. Λίγη το 116, εγκρίνεται. 117 ξεκινά, λίγη, εγκρίνεται. 118 με ε, προφορική τροπολογία της Κατερίνας Σολυνίβαν ξεκινά, κλείνει, εγκρίνεται 119 ξεκινά, λίγη, εγκρίνεται 120 ξεκινά, λίγη, απορρίπτεται 121 ξεκινά, λίγη, εγκρίνεται 122 ξεκινά, λίγη, εγκρίνεται 123 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 124 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 125 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 126 ξεκινά λίγη απορρίπτεται 127 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 128 κάποιο σχόλιο χωρίς όμως ε, μικρόφωνο ψηφίζουμε την Κώστα ε, θα κατέπιπτε μόνο αν ήμασταν υπέρ της τροπολογίας Βεζιά 128 σε δύο μέρη πρώτο μέρος ξεκινά λίγη εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος ξεκινά, λίγη, εγκρίνεται. 129 ξεκινά, λίγη, εγκρίνεται. 130 ξεκινά, λίγη, εγκρίνεται. 131 ξεκινά, λίγη, εγκρίνεται. 132 ξεκινά, λίγη, εγκρίνεται. 133 133, όχι 134 λέει πρόεδρος, με συγχωρείτε. Ξεκινά. λίγοι, Εγκρίνεται. 134. Ξεκινά. λίγοι, Εγκρίνεται. 135. Ξεκινά. λίγοι, Εγκρίνεται. 136. Ξεκινά. Λίγη εγκρίνεται 137 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 138 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 139 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 140 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 141 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 142 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 143 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 144 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 145 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 146 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 147 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 148 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 149 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 150 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 151 χωριστά σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα ε, κλείνει εγκρίνεται δεύτερο μέρος ξεκινά λίγη απορρίπτεται 152 ξεκινά λίγη απορρίπτεται 153 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 154 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 155 θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε μαζί την 155 μέχρι 158. Ποιος είναι υπέρ των όχι μία-μία, 154 υπέρ ε, εγκρίνεται, 155 κλείνει, εγκρίνεται, 156 ξεκινά, κλείνει, εγκρίνεται, 157 ξεκινά, κλείνει, εγκρίνεται, 158 ξεκινά, κλείνει, εγκρίνεται, 159 αποσύρεται 160 ξεκινά κλείνει εγκρίνεται 161 ξεκινά κλείνει απορρίπτεται 162 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 153 ξεκινά κλείνει απορρίπτεται 164 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 165 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 166 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 167 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 168 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 169 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 170 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 171 ξεκινά Λίγη. Εγκρίνεται. 172. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 173. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. Ε, συμβιβαστική ε, ήττα. Ε, ξεκινά. Λίγη. Ε, εγκρίνεται. 174. Ξεκινά. Λίγη. Απορρίπτεται. 176 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 178 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 179 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 180 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 181 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 182 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 184 και μπαντία κούτσετ είναι ταυτόσιμες ξεκινά κλείνει εγκρίνονται Α, δεν, σε Επαναλαμβάνουμε την 184-185 ξεκινά Λίγοι εγκρίνονται. 186. Ξεκινά. Έχει καταπέσει, με συγχωρείτε. 187. Ξεκινά. Κλείνει. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 188. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 190. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 191. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 192. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 193. Ξεκινά. Λίγη εγκρίνεται 194 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 195 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 196 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 197 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα ξεκινά λίγη εγκρίνεται δεύτερο μέρος ξεκινά λίγη εγκρίνεται 198 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 197 99 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 200 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 2001 ξεκινά 201 με συγχωρείτε εγκρίνεται 202 εγκρίνεται 203 ξεκινά Λίγη. Εγκρίνεται. 204. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 1. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 2. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 3. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 4. Ξεκινά. Λίγη εγκρίνεται 8 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 9 ξεκινά λίγη απορρίπτεται 5 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 6 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 7 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 10 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 11 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 12 καταπίπτει η 13 η... κλείνει εγκρίνεται 14 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 15 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 16 ξεκινά. Λίγη. Απορρίπτεται. 18 ξεκινά. Κλείνει, εγκρίνεται. 19 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 20 ξεκινά. Λίγη εγκρίνεται 21 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 22 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 23 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 24 ξεκινά λίγη εγκρίνεται 25 ξεκινά λίγη απορρίπτεται 26 ξεκινά, λίγη, απορρίπτεται, 27, κλείνει, απορρίπτεται, 28, ξεκινά, λίγη, εγκρίνεται, 29, ξεκινά, λίγη, απορρίπτεται. Ερχόμαστε στην τελική ψηφοφορία. Ποιος είναι για τη συνολική έξοδο. Εσύ Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 31 ομόφωνα, ούτε η κυρία Μπεζίε βλέπω. Οπότε συγχαίρουμε τον κύριο Παπα-Νικολάου. Πολλές από τις τροπολογίες σας γίνανε αποδεκτές κυρία Μπεζία, λέει η πρόεδρος. Και τώρα ερχόμαστε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ δεν έχουμε πολλή δουλειά πια σήμερα διότι η έκθεση της κυρίας Ναβινταλόβα έχει ήδη τελειώσει και τώρα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο και τους συναδέλφους του της Ένωσης Λερον Κόντρ, οι συναντήσεις. Περί τίνος πρόκειται θα μας πούν ακριβώς οι κύριοι αυτοί. Δεν θα ήθελα τώρα να επισέλθω σε λεπτομέρειες γιατί νομίζω ότι εσείς πρέπει να παρουσιάσετε το ευαγιές έργο σας και γι' αυτό σας καλέσαμε. Θέλω λοιπόν τώρα Παρακαλώ όλους τους συναδέλφους να καθίσουν. Το ίδιο ισχύει και για τους βουλευτές. Η νεαρά στο βάθος της εσούσης, παρακαλώ. Η νεαρά με ε, τα γκρίζο μπορεί παρακαλώ να καθίσει κάτω δεν είναι δυνατόν. Είναι τρομερό. Τώρα λοιπόν η, η Ρονκόντρ. Κύριε Τροπεάνο, έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω εσάς αλλά και τους συναδέλφους σας της Επιτροπής σας για την πρόσκληση την οποία μας απευθύνατε και τον χρόνο ομιλίας που μας δίνετε. Δεξιά μου έχω την κυρία Οντίλ Φόβ, η οποία είναι υπεύθυνη ε, για πολιτιστικά θέματα ε, του Ολλανδικού Λιμπούρ. Θα ε, της δώσουμε βεβαίως τον λόγο, αλλά θα ήθελα επίσης να σας παρουσιάσω τον κύριο Ζωζεφ Ντίλεν σε ταμεία, τον κύριο Ολίβ Ουγιάτ, ο οποίος είναι σύμβουλος, τον Ρέινερ, ο οποίος εκπροσωπεί εδώ ε, τον δήμαρχο του Μανχάιμ και τον τελευταίο φίλο μας που είναι ο βοηθός ε, της Οντίλε Βόλφ. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω σύντομα το δίκτυό μας. Έστω και αν μερικοί μεταξύ μόνο το γνωρίζετε και μάλιστα είχατε και την ευκαιρία να εργαστείτε μαζί μας. Πρόκειται λοιπόν για ένα δίκτυο το οποίο ονομάζεται "le rencontre" οι συναντήσεις, και που ε, αφορά ένα δίκτυο όλων των ερετών που ε, ασχολούνται με πολιτιστικά θέματα ερετών σε κάθε επίπεδο, κοινότητες, δήμους, νομαρχίες, επαρχίες η βάση σκέψης και δράσης δεν είναι μονάχα η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι υποψήφιες χώρες, δηλαδή το σύνολο των χωρών που εμείς αποκαλούμε η Μεγάλη Ευρώπη. Θα κάνω μια σύντομη παρουσίαση και μετά ίσως έχουμε και την ευκαιρία να κάνουμε μια συνάντηση. Ασχολούμεθα με πολλά πράγματα. Ας πούμε, ε, προωθούμε ε, πολιτιστικά θέματα σε όλα τα ευρωπαϊκά επίπεδα. Ε, μία από τις ιδέες μας, για να μην πω η αιμονή μας, είναι η δικτύωση ε, για θέματα πολιτιστικά σε κάθε τόπο και σε κάθε κοινότητα. Θέλουμε επίσης να ενισχύσουμε τον ρόλο του ερετού που ασχολείται με πολιτιστικά θέματα ε, όπου και αν αυτός δραστηριοποιείται. Γιατί ίσως εδώ να είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά ε, σε άλλα επίπεδα είναι πολύ δύσκολο να υπεραμεινθεί κανείς των πολιτιστικών θεμάτων. Επίσης ε, πρέπει να σας πω ότι έχουμε πάνω από 150 εκπροσώπους σε εθνική σε οργανώσεις και σε διεθνείς οργανισμούς και αυτοί οι 150 άνθρωποι προσπαθούν να βελτιώσουν και την εικόνα της Ευρώπης και την εικόνα της πολιτιστικής Ευρώπης. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ε, σας γνωστοποιήσω το τι κάνουμε αλλά και να ζητήσω και τη βοήθειά σας κατά κάποιο τρόπο έτσι ώστε να γίνει λίγο πιο γνωστό το δίκτυό μας. Μέχρι τώρα το δίκτυο πρέπει να σας πω ότι δημιουργήθηκε το 1914 έχουμε ε, σαν τακτική δράση την οργάνωση σε όλη την Ευρώπη συναντήσεων με τους ερετούς, τους καλλιτέχνες, όσους ασχολούνται με τα πολιτιστικά, πάντα σε συνεργασία με την πόλη που μας υποδέχεται και πάντα σε συνεργασία με τους ερετούς που εκλέγονται στην περιφέρεια ε, στην οποία, την οποία επισκεφτόμαστε. Έχουμε επίσης παρουσία στι Ευρωπαϊκέ πολιτιστικέ πρωτεύουσε και νομίζω ότι είμαστε το μόνο δίκτυο που ήδη από το 1992, τότε που ήταν η Μαδρίτη, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, ε, ξεκινήσαμε τη συνεργασία αυτή. Είμαστε το μόνο δίκτυο, λέγω, το οποίο παρακολούθησε όλες τις πολιτιστικές πρωτεύουσες για μας ε, το σχέδιό μας ε, είναι μια δυνατότητα που έχουν ε, οι πόλεις να συνενώνονται, να σκέπτονται μαζί και να κάνουν σχέδια για το μέλλον. Οργανώνουμε επίσης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, συναντήσεις με τους εθνικούς ερετούς της προεδρεύουσας χώρας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι τοπικοί αιρετοί να κατανοούν τι σημαίνει για έξι μήνες η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα λοιπόν αυτή την περίοδο είμαστε στην Ισπανία, είμαστε στην Μαδρίτη και ε, μετά από αίτημα των ερετών ε, οργανώνουμε διάφορες θεματικές συζητήσεις. Ε, θέματα τα οποία οργανώνονται είτε μονοθεματικά είτε εγκάρσια. Πάντοτε καλούμε όσους επαγγελματικά ασχολούνται με τον πολιτισμό ε, και θέλουμε να βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί. Τους δίνουμε την δυνατότητα λοιπόν να συναντώνται για να ανταλλάσσουν απόψεις. Πιστεύω λοιπόν ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις αντιπροσωπεύουν μια μοναδική ευκαιρία ε, και για τους πολιτικούς που ασχολούνται με τα πολιτιστικά θέματα αλλά και τους επαγγελματίες ε, του ε, πολιτισμού και δίνουν, δίνεται η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων, δίνεται η δυνατότητα οι μεν να γνωρίσουν τα προβλήματα των δε, να δουν οι χώρες πώς οι άλλες χώρες αντιμετωπίζουν και λύνουν ενδεχομένως κάποια προβλήματα. Πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα καταφέρουμε να επιτύχουμε αυτό το δικαίωμα στον πολιτισμό που πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με το δίκτυό μας πιστεύω ότι δημιουργούμε δυνατότητες, ανοίγουμε ορίζοντες, διότι ο πολιτισμός είναι καταλήτης για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καταλήτης για το μέλλον. Δεν θα αναφερθώ εδώ στη σχέση ανάμεσα ε, στην κοινωνία, την οικονομία και τον πολιτισμό. Ε, εγώ απλώς θέλω να σας πω ότι προσπαθούμε να είμαστε ανοιχτοί ε, μέσω του πολιτισμού σε όλες τις δραστηριότητες των τοπικών και κοινωνιών. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ σε μια πρωτοβουλία. Πριν από μερικά χρόνια δημιουργήσαμε ε, και δημοσιεύσαμε μια πράσινη βίβλο της πολιτιστικής ε, πολιτικής και στρατηγικής στην Ευρώπη και τώρα εκπονούμε και είμαστε έτοιμοι να δημοσιεύσουμε την Λευκή Βίβλο. Το έγγραφο αυτό δεν θέλουμε να δημοσιευθεί στην παραδοσιακή μορφή ενός έργου. Θέλουμε να το παρουσιάσουμε στο ίντερνετ ε, με διαδραστική ε, και βαθμιαία ε, μορφή έτσι ώστε όσοι ασχολούνται με τον πολιτισμό, εκλεγμένοι ή επαγγελματίες να είναι σε θέση να το επισκεφθούν, να το διαβάσουν. Πιστεύουμε ότι και μετά την κρίση αλλά και στη διάρκεια της κρίσης που περνάμε ε, θα πρέπει να ξανασκεφτούμε κάποια πράγματα έτσι ώστε να βρούμε μια νέα στρατηγική, ένα νέο στάδιο. Πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τους διανοητές, πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τους ανθρώπους του πολιτισμού έτσι ώστε μαζί να σκιαγραφίσουμε τις νέες περιόδους που ανοίγονται μπροστά μας και για, κατά αυτή την έννοια θα ήθελα να σας ζητήσω να παρακολουθήσετε την, ε, τις εργασίες μας. Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Βόλφ. Κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε που μας προσκαλέσατε να έρθουμε εδώ και να σας εξηγήσουμε ποια είναι τα θετικά του να συμμετέχει κανείς σε αυτό το πολιτιστικό δίκτυο βεβαίω. και εγώ περιορίζομαι να σας μιλήσω για το ποια είναι τα θετικά για το Ολυμβούργο αλλά είμαι βέβαιος ότι και άλλα μέλη της Ρανκόντορ θα σας πούν τα ίδια. Η επαρχία μας, όπως ξέρετε, βρίσκεται στα νοτιοανατολικά των κάτω χωρών και 80% ε, συνορεύουμε με Βέλγιο και Γερμανία και μόνο 20% με την μητέρα χώρα, με την ε, Ολλανδία ακριβώ λόγω ε, αυτής της γεωγραφικής της τοποθέτησης η επαρχία μας έχει διεθνείς επαφές εκφύσεως ούτως Οπότε γι' αυτό και συνεργαζόμαστε στενά πάνω από 30 χρόνια. Και έχουμε επίσης έχουμε και επαφές και για, τη, για, για κάποια γλωσσικά θέματα, για κάποιες του πηγές, οπότε γι' αυτό τότε που γεννήθηκε το ευρώ με τη συνθήκη του Μαστρίχτ, από τότε ε, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε η Ευρώπη σε σμίγνη, σε μινιατούρα. Οπότε μπορείτε να έρθετε και να δείτε σε μια μέρα όλη την Ευρώπη μέσα από την επαρχία μας. Γι' αυτό μπορείτε να καταλάβετε τόσο, τόσο πολλά χρόνια χρειάζεται να ανταλλάξουμε εμπειρίες με την υπόλοιπη Ευρώπη για να μπορέσουμε να ε, δούμε ποια θα είναι η, η στάση, η νοοτροπία σε σχέση με την άρση κάποιων ε, φραγμών συνοριακών. Ε, τέρμα στα σύνορα για να μπορέσουμε αυτή μας η εμπειρία και η γνώση να την έχουν και άλλοι αλλά και εμείς να ακούσουμε του άλλους και έτσι όλοι μαζί να βελτιωθούμε και αυτό γίνεται σε ετήσια βάση και όσον αφορά την ε, ε, πολιτιστική μας πολιτική οπότε αυτό θεωρήσαμε ότι είναι κάτι που πρέπει να γίνεται σε καθημερινή βάση σαν Επαφέ για αυτή τη διαδικασία. Είπαμε ότι δεν θα αφήσουμε τα πράγματα στην τύχη. Πρώτα-πρώτα κάναμε ε, έναν κατάλογο από τα πολιτιστικά ευρωπαϊκά δίκτυα. Τα περισσότερα από αυτά είναι μια πλατφόρμα για πολιτιστικά ιδρύματα και άλλα τέτοια ε, δίκτυα επικεντρώνουν την δράση τους σε αστικές περιοχές ή στην ε, Ήπεθρο. Αφού κάτσαμε και αναλύσαμε το τι γίνεται με τους ειδικού τελικά Διαλέξαμε να ενταχθούμε στον φορέα Λέραν Κόντρα για πολλούς λόγους. Κατά τη γνώμη μας πρώτα-πρώτα είναι το μόνο δίκτυο το οποίο συνενώνει τις πόλεις, την ε, Ήπεθρο αλλά και κάποιες περιφερειακές αρχές όπως πρόκειται και στην περίπτωση τη δική μας, το Λιμβούργο. Πρόκειται για ένα δίκτυο το οποίο συνενώνει ε, διάφορα στοιχεία, διάφορους φορείς πολιτιστικού, διαφόρων ε, επιπέδων διακυβέρνηση ούτω ώστε να υπάρχει ανταλλαγή ιδεών, γνώσεων και εμπειριών. Επίσης, έχει μέλη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και στις απότερε γωνιές της. Αυτό δίνει περισσότερο ενδιαφέρον, περισσότερες ε, ακούγονται, περισσότερη προβολή και επομένως έτσι ο ένας μπορεί να ενισχύσει τον άλλο και είναι δυνατόν κανείς να βρει τη θέση του στο ευρωπαϊκό και εθνικό στερεώμα. Επίσης, οι συναντήσεις των Ρανκόντρα αφορούν θέματα ευρωπαϊκά ε, στον πολιτικό τομέα. Οπότε, φέτος ας πούμε η Προεδρία έχει κηρύξει το έτος της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης, κάθε χρόνο συζητιέται το θέμα της πολιτικής πρωτεύουσας, οπότε ε, πάντοτε τα μέλη των Ρανκόντρ είναι ενημερωμένα για τις πολιτικές κάθε ε, συγκυρίας. Και ε, έχουμε ανανέωση, έχουμε περισσότερους που έρχονται στις συναντήσεις, οπότε έτσι η απόδοση της ευκαιρίας του δικτύου αυτού πολλαπλασιάζεται. Και με αυτή την προσέγγιση όποιος συμμετέχει μπορεί να διαλέξει σε ποια συνάντηση θα πάει ανάλογα με το περιεχόμενο. Αυτό παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι σε κάθε συνάντηση έχουμε κάποιους που ενδιαφέρονται για το ίδιο θέμα. Γενικώ, σε αυτόν τον τρόπο επίσης έχουμε κίνητρα για αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν και πάντοτε ε, οι συναντήσεις μας αφορούν κάποιες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε οπότε όλοι όσοι συμμετέχουν εισφέρουν την εμπειρία τους ε, και όλοι εποφελούνται. Βεβαίως κυρίε και κύριοι, δεν θέλω να σας κρύψω ότι η Εουρέγιο και το Μάστριχτ ε, αφορούν το ότι διαλέξαν ποια ήταν η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα για το 2018, κάτι το οποίο βοήθησε στις επιλογές μας. Ε, εμείς συμφωνούμε με τις επιλογές αυτές και δεν νομίζουμε ότι υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό το να ε, χρησιμοποιήσει κανείς την ποιότητα του μέλους για να πετύχει περισσότερη ποιότητα, καλύτερο περιεχόμενο και έτσι κι αλλιώς ε, το θέμα είναι να πετύχουμε το στόχο μας μέσω του, του, να ανταλλάξουμε εμπειρίες και νομίζω ότι ξεκαθαρίστηκε το ότι ε, τελικά αυτό το οποίο θέλουμε είναι όχι απλώς να προωθήσουμε την, ε, το, το σαν πρωτεύουσα πολιτιστική, πολύ περισσότερα πράγματα. Γι' αυτό και έχουμε την Φλωριάντ, αυτήν την ε, έκθεση για τα λουλούδια 2012, έχουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίου 2012, επίσης έχουμε το Μανιφέστα σε συνεργασία ε, με το Βελγικό Λιμβούργο που είναι μια διεθνή εκδήλωση τέχνη. Οπότε γι' αυτό και κανεί καταλαβαίνει το προβλαστικό αποτέλεσμα των ε, ε, δικτύων και όλα αυτά τα οποία μα ενώνουν στην Ευρώπη, όλα αυτά που έχουμε κοινά. Επομένω θέλουμε μια καλύτερη Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο. Να βρούμε ποια είναι τα κοινά μα, να βρούμε ε, τι, τι ανταλλαγέ υπάρχουν μεταξύ των διαφορών εθνών και αυτό βέβαια γίνεται με μικρά βήματα, βαθμία ε, καλύτερα είναι αυτά τα πολλά μικρά βήματα παρά το μεγάλο άλμα. Ε, γι' αυτό θεωρούμε ότι το δίκτυο Rancontr ε, το οποίο αποκλείει το να αφήσει κάποιον απ' έξω. Είτε αυτό είναι η ύπεθρος, είτε αυτό είναι η πόλη, είτε αυτό είναι οι περιφερειακές αρχές. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθεια όσον αφορά την πολιτική συνεργασία και έτσι πρόκειται και όσον αφορά την εμφάνιση και όσον αφορά το περιεχόμενο να έχουμε εξελίξεις ενδιαφέρουσες και σταθερή πρόοδο. Οπότε, αυτό σημαίνει ε, συνάντηση και λέει σε πάρα πολλές ε, γλώσσες την ίδια λέξη ομιλήτρια περί αυτού πρόκειται, συνάντηση ε, θα ήθελα τώρα κάτι να σας πω, ε, εν κατακλείδη. Ε, μισό να σας δώσω το λόγο. Συνεχίζει ο μιλητής γιατί θέλουμε να σας καλέσουμε σε όλες μας τις εκδηλώσεις. Ε, αυτό πρώτον και δεύτερον, όλοι οι, οι αιρετοί στην Ευρώπη να ξέρετε ότι προσέχουν τις εργασίες της Ευρωπαϊκής ε, Κοινοβουλικής σας Επιτροπής και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, θεωρούμε ότι έτσι θα βγουν οι καθυντήριες γραμμές, οι προοπτικές για την πολιτιστική Ευρώπη που όλοι ποθούμε. Εμείς σας ευχαριστούμε. Λεπρόντος και συνεχίζω στα... Ευχαριστώ όταν είμαι σε αυτή τη θέση έχω συνεργαστεί με τη Ρονκόντρο σε διάφορα θέματα οπότε ξέρω τι κάνετε δεν ξέρω αν ξέρετε εσείς τι κάνουμε σχετικά με την πολιτιστική ε, πολιτική και ε, τι γίνεται. Έχουμε απευθύνει από πέρυσι το φθινόπωρο μία, ένα ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον πολιτισμό και την περιφέρεια οπότε και εσείς θα έπρεπε να κοιτάξετε να επηρεάσετε την Επιτροπή του ε, θέματος αυτού διότι νομίζω ότι έχετε λάβει 250.000 ευρώ από τον κοινοτικό Κορβανά είναι 16% του προπολογισμού σας ίσως για άλλους δεν είναι πολλά αλλά δεν είναι ένα μικρό ποσό οπότε ε, ε, εφόσον ετοιμάζει βάζετε μία λευκή βίβλο την οποία έχετε δημοσιεύσει θα έλεγα να την ε, συνδυάσετε με ε, την ε, προφορική μας επερώτηση από ε, πέρυσι το φθινόπωρο διότι χρειαζόμαστε βοήθεια σε αυτό το τομέα. Βεβαίως ελέγχθη ότι και η Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο συνεργάζεται στον τομέα αυτό και εγώ προέρχομαι από μία περιοχή όπου επίσης εμπλέκεται ή στον πολιτιστικό τομέα οπότε αυτά τα οποία κάνετε τα θεωρώ πολύ σημαντικά και αντιλαμβάνουμε ότι η επόμενη συνάντησή σας θα γίνει στην Κροατία στη Γέκα μια ωραία εποχή οπότε έχετε σκεφτεί ίσως να κάνετε κάτι στην πρώην δημοκρατία της Μακεδονίας ή στο Σεράγιο ή στο Νόβισαντ για γιατί και αυτές οι χώρες ε, θα είναι ή είναι ήδη υποψήφιες για ένταξη για να περιληφθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οπότε ε, θα έπρεπε ίσως να περιλάβετε και την Αλβανία ε, έχετε πάει στη Βενετία οπότε δεν, θα πάτε στη Βενετία δεν είναι τόσο μακριά οι περιοχές αυτές θα έπρεπε ίσως να προωθηθείτε προς αυτές τις χώρες γιατί χρειάζονται βοήθεια καθότι δεν υπάρχουν καμία βοήθεια από τα κράτη αυτά για τις περιφέρειες και καλό θα ήταν να έρθετε σε επαφή με τους τοπικούς εκπροσώπους κατά να μπορέσουν να επιτύχουν κάτι καλύτερο στον τομέα που σας απασχολεί με τη δικιά σας όθηση. Η κυρία Νεβενταλόβα από τη Σλοβακία έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ να σας ευχαριστήσω για το έργο το οποίο επιτελείται, μια που είπαμε τόσα πολλά. Αλλά δεν κάναμε τόσα πολλά για τον πολιτισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένω, γι' αυτό και θα πρέπει οι προσπάθειές μας να συντονιστούν. Τώρα, θέλω να ρωτήσω τα εξή. Είπαμε τι θα κάνουμε με τις τρίτες χώρες, ε, πρέπει να υπάρξει συνεργασία και εκτός Ευρώπης. Άλλες μεσογειακές χώρες ε, ενδεχομένως. Εγώ είχα κάποιες σχετικές επαφές με το Τατζικιστάν. Γιατί πρέπει να κατευθυνθούμε και στο παλιό Σοβιετικό μπλοκ, γιατί ξέρετε ότι σε εκείνες τις χώρες ε, υπάρχει ακόμα θέμα. Ε, θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια από τα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης όσον αφορά τους νέους. Δεν προσέχουν τόσο πολύ την πολιτική ε, ε, ζωή εκεί πέρα. Οι νέοι ασχολούνται κυρίως με το κομπιούτερ, με το ίντερνετ. Άρα, να στραφούν προς τα εκεί, προς τους νέους, στις πρώην σοβιτικές δημοκρατίες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόρις από την Πολωνία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για αυτή την Υπάρχει ιδιαίτερος λόγος στον τομέα αυτό, ιδίως όσον αφορά το νέο προϋπολογισμό και την ε, ε, ατζέντα για το 2014 έως 2020. διότι υπάρχουν δυνατότητες στην ε, νέα δημοσιονομική πολιτική. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τη μετάφραση, λέει η πρόεδρος. Παρακαλώ τη γερμανική καμπίνα να μπορέσει να πατήσει κάποιο κουμπί γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν, ακούγομαι, δεν ακούγεται η μετάφραση. Ε, ο κύριος ακούγεται, όχι όμως οι κυρίες. Λοιπόν, ε, θα ε, υπάρξει συνεργασία και στα πλαίσια της ανατολικής συνεργασίας και της Μεσογείου γιατί και εκεί προβλέπονται πολιτιστικές κινήσεις. Το θέμα με την συνεργασία με την Επιτροπή Περιφερειών ήταν ένα που ήθελα και εγώ να θίξω διότι προηγουμένως αναφέρατε ότι θα έπρεπε να έρθετε σε επαφή με τις πολιτιστικές πρωτεύουσες. Αντιλαμβάνομαι ότι σήμερα το απόγευμα θα είστε σε μία εκδήλωση, αλλά τι είναι αυτή η συνεργασία, διότι ξέρω ότι οι 18 πόλεις της Γερμανίας και οι 11 της Ουγγαρίας έχουν δημιουργήσει ένα δίκτυο και συνεργάζονται στενά. Δεν ξέρω αν εσείς ε, εργάζετε εκ του παραλίου ασύλου ή έχετε ενταχθεί επίσης. Θα ήθελα να ξέρω πώς γίνεται η δικτύωση με το πολιτιστικό αυτό σύνολο. Θα παρακαλούσα λοιπόν τώρα να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα, οι συνεργασίες τις οποίες έχουμε με άλλες ε, πόλεις και άλλες ε, χώρες ανατρέχουν στην γένεση του δικτύου μας. Δηλαδή ευρύτερη Ευρώπη είναι η ύλη μας. Έχουν πάει Σερβία, Σκόπια, το Σαράγιβο, Βοσνία, Σαρζεγοβίνης, όλες αυτές οι πόλεις και οι περιοχές είναι στο δίκτυο, οπότε έχουμε με όλους αυτούς ε, στενούς δεσμούς και συνεχώς κανονίζουμε επαφές, ώστε να υπάρχει διάλογος και αμοιβαίο feedback. Οπότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μην υπάρχει βέβαια και μεγάλη κατάτμιση των ε, προσπαθειών, να δούμε τι θα γίνει και με τη Μεσόγειο και πάντα να πρετανεύει το πνεύμα το ότι η δουλειά μας να αφορά το τι γίνεται όσον αφορά τη συλλογική, δαφική προσπάθεια, να μην έχουμε επικάλυψη με άλλα δίκτυα τα οποία δουλεύουν σε άλλο επίπεδο ε, θεσμικό, καλλιτεχνικό, γιατί για μας αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να έχουμε στενές σχέσεις με κάποια δίκτυα τα οποία να παρομοιάζουν με το δικό μας και να δρουν στην ε, ήπειρό μας. Έχουμε αυτό που λένε interlocal. Αυτό το δίκτυο αφορά κάποιες ε, ισπανοαμερικανικές, δηλαδή νότιοαμερικάνικους φορείς. Έχουμε σχέσεις με αυτό το δίκτυο και αυτό το οποίο θέλουμε στα πλαίσια της ε, ομάδας εργασίας σε ΖΕΛΗ να πρώτα-πρώτα έχουμε διάλογο, ή κοινέ δράσει με τέτοια δίκτυα που μοιάζουν το δικό μα σε άλλε υπήρου, τόσο ώστε να υπάρχει ένα πάγιο διάλογο τη Ευρώπη μα με τον πολιτισμό άλλων υπήρων. Επίση, όσον αφορά την Πολωνία πιο συγκεκριμένα, πρόκειται να έχουμε παρουσία στη χώρα αυτή με την ευκαιρία τη Προεδρία που θα αναλάβει η χώρα αυτή του χρόνου και θα συνεχίσουμε τη δουλειά μα με πόλει πολωνικέ. Όσον αφορά δε τι περιφέρειες Βεβαίως και η Επιτροπή των Περιφερειών ε, είναι συνεργάτης ε, βασικός και τους προσκαλούμε στις ε, συναντήσεις μας και βέβαια όσο επιτρέπει όσο επιτρέπουν του καθενός όσον αφορά τώρα την πολιτική πρωτεύουσα βεβαίως όπως τα είπε η συνάδελφος προσπαθούμε να δούμε το ότι πολλές φορές υπάρχει ενδιαφέρον να αναλυφθεί ένα τέτοιο έργο σε σχέση με ε, την ανάληψη του, του ρόλου της πολιτικής ε, πρωτεύουσας. ας πούμε ε, το παράδειγμα της Μαδρίτης θα καλέσουμε όλους τους εκπροσώπους των πόλεων που ήταν υποψήφιες πόλεις Ισπανούς, Πολωνούς, Μαδρίτης δηλαδή και Πολωνίας γιατί θεωρούμε ότι άπαξ και έχει επιλεγεί μια πόλη εκπροσωπεί όλες τις πόλεις της χώρας επομένως όλοι θα πρέπει να ε, κληθούν και επομένως γι' αυτό και παρακολουθούμε το έργο της Επιτροπής σας αλλά και την έκθεση ε, ΠΡΕΤ που αφορά τις πολιτικές πρωτεύουσες. Πάντως, να, αν γίνεται να έχουμε πιο στενή συνεργασία επί τη βάση περιφερειών, συγκεκριμένων περιοχών και εμείς ε, πρώτη θέμεθα να έχουμε συγκεκριμένη συνεργασία και στενή συνεργασία με την ε, κοινοβουλευτική σας επιτροπή. Γιατί η Ευρώπη και ο πολιτισμός σημαίνει και ε, περιφέρεια. Συνεχίζει στα Ολλανδικά η κυρία Βόλφς. Κυρία Πρόεδρε. Το βασικό πλεονέκτημα του, του, του δικτύου Rancontr είναι ότι είναι ένα δίκτυο στο οποίο ανήκουν κάποιες πόλεις που έχουν διατελέσει πολιτικές πρωτεύουσες και κάποιες άλλες που φιλοδοξούν να είναι. Και αυτό φράγει τη θεματική μας, γιατί πρόσφατα ασχοληθήκαμε με τις επιπτώσεις της ε, κρίσης, της οικονομικής, πάνω στην ε, πολιτιστική πολιτική. Επομένως πρέπει να δούμε πώς θα βρούμε σπόνσορες και χορηγούς εκτός κρατικών φορέων γιατί έχοντας συνεργασία και ανταλλαγές μεταξύ αυτών των πόλεων που σας ανέφερα έχουν προσταμένη αξία διότι ακριβώς οι υποψήφιες πόλεις μπορούν η μία να διδάξει στην άλλη πολλά. Το Έσεν, η Κολονία είναι τέτοιες περιπτώσεις που μετέχουν στο γερμανικό κομμάτι του δικτύου. Οπότε ασχολούνται με όλα αυτά τα συγκεκριμένα θέματα, ανταλλάσσουν πληροφορίε, ανταλλάσσουν γνώσει, εμπειρίε σε σχέση με το τι πάει να πει να είναι κανεί πολιστική πρωτεύουσα. Πώ οργανώνονται τα πράγματα κλπ. Και στη δική μα την επαρχία, ξέρετε, έχουμε κάποιου φορεί που συμμετέχουν σε προγράμματα και στο εξωτερικό. Οπότε, για να δούμε τώρα, όσον αφορά εκείνη σα την, ε, την ερώτηση για Λετωνία, Εστονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Ανατολική Ευρώπη, όλες αυτές οι χώρες είναι στο Ρανκόντρο. Ναι, αλλά βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι χώρες αυτές. Είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεω. Η Μαρή Τερέζ Ευχαριστώ. Σε συνέχεια τον όσων είπε η Κατερίνα, μίλησαμε χθε για την έκθεση Μπαδία. Ακριβώ για να μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε του νέου. Για να δούμε πώ. Όσον αφορά αυτού του φορεί, του πολιτιστικού, ε, αν μπορείτε και να, να μας πείτε συνάδελφε τι γίνεται όσον αφορά την δημιουργία, την καλλιτεχνική, την πολιτιστική γενικότερα. Ε, σας ευχαριστούμε, αλλά ε, νομίζω ότι τώρα μας βάζετε πολύ ψηλά τον πύχη και, και, και, τη φιλοδοξία, γιατί όπως είπε και η Πρόεδρος υπάρχουν και κάποιοι όρια στη δράση μας, γιατί να σταθώ στο θέμα αυτού του οράματος, αυτού του, του, αυτής της ιδέας για την καλλιτεχνική παιδεία και εκπαίδευση. Ξεκινήσαμε μόλις πέρσι στο Βίλνιους τον προβληματισμό. Τότε ήταν ε, πολιτική πρωτεύουσα το Βίλνιους και καλέσαμε εκπροσώπους των δικτύων που ασχολούνται με αυτό και ήρθαν και οι δικοί μας βέβαια, οπότε ξεκίνησε η υπόθεση αυτή. Ε, ξέρετε, δεν εξαρτάται από εμάς να αναλάβουμε δράση. Παιδαγωγική είναι η δράση μας, όπως είπα. Στο δίκτυο θέλουμε να μπορέσουμε και να βοηθήσουμε να προχωρήσουν κάποια μικρά προγράμματα στην Ευρώπη που θα γινόντουσαν μόνο εάν βοηθήσουν τέτοιοι φορείς για τη δημιουργία, μετάφραση, τους καλλιτέχνες. Ενημέρωση, επομένως, παιδαγωγική δράση με δίκτυα, γιατί πρόκειται για πολύ σημαντικό τομέα, θεωρούμε. Η παιδεία και εκπαίδευση καλλιτεχνική. Πάντως θα θέλετε να δείτε τι έγινε ε, στο Βίλνιος ακριβώς. Υπάρχουν αυτά στο website που έχει το Rancontre στα γαλλικά. Κυρία Πακ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε που ήρθατε να μα δείτε, καλή συνέχεια. Οπότε θα, δείτε κι εσείς και εμείς τι, τι θα κάνουμε και θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε, να συνεχίσουμε αυτή τη διαδρομή για ε, τα πολιτιστικά στις περιφέρειες και δεν ξέρω που πάμε <laughs> αλλά οπωσδήποτε ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα αγγίξουν, θα ευαισθητοποιήσουμε την Κομισιόν στα γερμανικά. Τώρα έχουμε το σημείο 12 της συνεδρίασης των συντονιστών. Δεν ήμουν παρούσα, αλλά νομίζω ότι λάβατε όλες τις ενημερώσεις στο στο email σας εγώ θέλω να μιλήσω πρόεδρε για αυτό το σχέδιο ψηφίσματος Δεν είχαμε το χρόνο για να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Μήπως γίνεται ε, να έχουμε καμιά μερούλα παραπάνω για να ασχοληθούμε με την ε, ουσία του θέματος και τις ε, τροπολογίες. Δεν ξέρω τι λένε συνάδελφοι, αλλά πρόκειται για αυτό που το συζητήσαμε χτες. Μήπως γίνεται να έχουμε την ευκαιρία κάπως να το συζητήσουμε. Εχθές το βράδυ συμφωνήσαμε ότι μετά από σήμερα αυτό επρόκειτο να ε, μοιραστεί. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, ο Ήβο. Ευχαριστώ. Ε, ούτως ή άλλως ε, έχει μοιραστεί από την προηγούμενη Πέμπτη. Ίσως εσείς να το λάβατε αργότερα κύριε Μπαντία, δεν ξέρω. Ε, το θέμα είναι να μου πείτε ποιο είναι υπεύθυνο για το θέμα αυτό στην ομάδα σας, ε, να έρθω σε επαφή μαζί του και να συζητήσω το θέμα, γιατί βεβαίω είμαστε απολύτω ανοιχτοί. Είστε εδώ σήμερα. Θα προσπαθήσω να βρω μια λύση σήμερα. Λοιπόν, θα το διευκρινίσουμε ε, διμερός μεταξύ της κυρίας Μπέλετ και του Ήβο και μετά θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο θέμα play agents. Δεν νομίζω ότι έχουμε άλλα προβλήματα Ήβο. Αυτή είναι μία αίτηση της Doris Πακ, όχι εν ονόματι ε, της, ε, ε, της, ε, της Επιτροπής. Ήταν μία πρόταση του ΕΛΚ την οποία, η οποία έγινε αποδεκτή από τους συντονιστές και περνάει σαν πρόταση της ε, Επιτροπής. Άρα τελειώνει η συνεδρίαση και πιστεύω ότι έχετε πολλά να κάνετε στο γραφείο σας. Σας ευχαριστώ.